μυαλό μας. Καλωσορίσατε λοιπόν και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Βαν Όρντεν. Ακόμα ένα θερμό χαιρετισμό προ του εκπροσώπου του Ινδικού Κοινοβουλίου. Θα είστε πάντα πρόσδεκτοι στην Ευρώπη. Και τώρα για να κλείσουμε τη σημερινή συζήτηση για τι δηλώσει ε, στην προετοιμασία του Συνόδου Κορυφή 25 και 26 Ιουνίου θα δώσω το λόγο πρώτα στον πρόεδρο, αντιπρόεδρο τη Επιτροπή κύριο Τίμερμαν. Ευχαριστώ. Να απαντήσω σε ορισμένα από τα σχόλια τα οποία έχουν γίνει. Για την Ελλάδα πρώτα. Επιμένω ότι η Κομισιόν θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για την εξέβρεση μιας συμβαστικής λύσης που να είναι αποδεκτή για όλους και η οποία βασίζεται στην ιδέα ότι δεν πρέπει να αφήσουμε τον ελληνικό λαό να βασανίζεται περισσότερο και θα πρέπει να βρούμε μια λύση στα προβλήματά του. Αυτοί από εσά οι οποίοι επιχειρηματολογήσαν, όπως ο κύριος Νάτελ και η κυρία Λεπέν, ότι είναι φίλοι του ελληνικού λαού και είναι εναντίον του ευρώ και πιστεύουν ότι η Ελλάδα θα πρέπει να φύγει από το ευρώ, θα πρέπει να αλλάξουν θέση ή να ξανασκεφτούν αν είναι πράγματι φίλοι της Ελλάδας. Γιατί η ευρεία πλειοψηφία των Ελλήνων θέλει μια λύση μέσα στο ευρώ. Δεν θέλουν να φύγουν από το ευρώ. Αν είσαστε τόσο μεγάλος φίλος Ελληνικού λαού, μήπω μήπως θα πρέπει να ακολουθήσετε την άποψη των Ελλήνων για το θέμα αυτό. κάποιος δίπλα στην κυρία ε, Λεπέν κάνει ένα ανέβμα σαν να είναι τελείως παραλογισμός όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Εν πάση περιπτώσει με τέτοιους φίλους εγώ προτιμώ τους εχθρούς μου λέει ο κύριος Τιμέρμανς. Ένα άλλο σημείο που με εντυπωσίασε είναι ότι ο κύριος Νάτελ διαμαρτυρήθηκε για το γεγονός ότι οι βουλευτές του δεν μπορούσαν να έρθουν χθε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λόγω μιας απεργίας. Μα εγώ νόμιζα ότι <laughs> το κόμμα το έκανε ό,τι μπορούσε για να ξεφορτωθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν μπορείτε να τα έχετε όλα κύριε Νάτελ. Ελπίζω λοιπόν ότι οι Βρετανοί βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν θα ξεχάσουν την κληρονομιά τους στην κοινοβουλευτική ότι είναι ανοιχτή προς τον κόσμο και ότι έχουν αρκετή εμπιστοσύνη στον εαυτό τους ώστε να μην σκεφτούν να κάνουν τύχη με, στα όρια της Ευρώπης. Και αυτό με φέρνει στο δεύτερο σημείο που είναι το θέμα της μετανάστευσης. Ή θα βρούμε ευρωπαϊκές λύσεις ή δεν θα βρούμε καθόλου λύσεις που να αντιμετωπίσουμε μας προβλήματα. Αυτή είναι η βαθιά μου πεποίθηση. Νομίζω ότι το να δίνουμε την εντύπωση ότι με το να κρατάτε τους ανθρώπους έξω από την Ευρώπη θα λύσετε το πρόβλημά σας, αυτό δεν είναι μονάχα ηθικά ύποπτο, είναι πολιτικά ανέφικτο. Δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν είμαστε η Αυστραλία, δεν είμαστε περιστοιχιζόμενοι από ένα ωκεανό. Δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιες λύσεις. Και τι θα πείτε σε μια οικογένεια που ξεφεύγει από πολέμους στην ε, Δαμασκό ή στην, ε, σε άλλες περιοχές στη Λιβύη. Θα τους πείτε δεν σας δίνουμε άσυλο, μείνετε εκεί πέρα να σκοτωθείτε, μείνετε στην πατρίδα σας να σκοτωθείτε. Ναι. Πήγαινε να το πείτε σε χώρε όπω είναι η Ιορδανία. Πήγαινε να το πείτε σε χώρε όπω το Λίβανο, όπω ο Λίβανο που έχει το 1 τέταρτο του πληθυσμού του να είναι πρόσφυγε. Καιρό να ξανασκεφτούμε αυτήν την ιδέα ότι με το να κρατάμε έξω από τα όρια τη Ευρώπη του πρόσφυγε θα λύσουμε τα προβλήματα αυτά. Η Ευρώπη πρέπει να βρει μια βιώσιμη λύση που να βασίζεται στι αξίε μα. Αν εμεί χάσουμε τι αξίε μα για αυτό το θέμα, θα τι χάσουμε και για όλα τα άλλα θέματα. Πρέπει να το κάνουμε και να διατηρήσουμε τι αξίε μα για όλα τα θέματα και τα θέματα που έχουν να κάνουν με τους πολίτες μας. Ζητώ λοιπόν από το Συμβούλιο αύριο να ακολουθήσει τη λογική τη Κομισιόν. Δώστε μα καλύτερε λύσει, καλύτερα επιχειρήματα ή δεχτείτε τι προτάσει μα. Η Κομισιόν θα παραμείνει πιστή στην πρότασή τη και αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου πιστεύω ότι με υποστηρίζει και μου δίνει λόγο να παραμείνω πιστό στη θέση τη Κομισιόν. Προσπαθήσαμε θελοντικά συστήματα, απέτυχαν στο παρελθόν. Και εδώ είναι ένα θέμα πολιτικής και ηθικής ακαιρεότητας να το καταλάβουμε και να αντλήσουμε τα απαραίτητα συμπεράσματα. Ελπίζω λοιπόν ότι τα μέλη του Συμβουλίου θα εμπνευστούν από αυτή τη συζήτηση αν πάρουν το θέμα αυτό σοβαρά. Για αυτό που είπε ο κύριος Φερχόφστατ για την Ουγγαρία. Η Κομισιόν είναι σε στενή διαβούλευση με την κυβέρνηση της Ουγγαρίας. Ποιοι είναι οι τεχνικοί λόγοι που οδηγούν σε αυτήν την απόφαση κτλ. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει πράγματι αναστολή, είναι απλώ ίσω μόνο φήμε. Προσπαθούμε να διακριβώσουμε τι ακριβώ γίνεται. Προφανώ θα ζητήσουμε από όλα τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν του κανόνε και αν υπάρχει μια έκτακτη κατάσταση υπάρχουν ενδείξει ότι η Ουγγαρία αντιμετωπίζει ένα τεράστιο ρεύμα προσφύγων. Υπάρχουν σε αυτή την περίπτωση εργαλεία, σε αυτή την περίπτωση να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση ακραίου χαρακτήρα, αλλά το να σταματήσουμε απλώ την είσοδο των προσφύγων δεν είναι ένα από τα εργαλεία που επιτρέπονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα βοηθήσουμε όλα τα κράτη-μέλη και συγκεκριμένα την Ουγγαρία. Εμεί συζητούμε μαζί του για το θέμα αυτό, αλλά παροτρύνουμε όλα τα κράτη-μέλη <clears throat> να σεβαστούν του κανόνε που έχουμε από κοινού συμφωνήσει. Και θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε αυτή, να παρακολουθούμε αυτή την κατάσταση στην Ουγγαρία. Εν τέλει, εν τέλει κύριε Πρόεδρε. Θέλω να τονίσω και πάλι εξ ονόματο τη Κομισιόν ότι αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο πρέπει να, πάρει, να κάνει τολμηρά βήματα προς τα εμπρός σε σχέση με το θέμα της μετανάστευσης. Αν δεν αποφασίσουμε τώρα θα πεθάνουν και άλλοι και δεν θα μπορέσουμε <clears throat> ποτέ να εφαρμόσουμε τους κανόνες αυτούς και τα απαραίτητα μέτρα που θα πρέπει από τον Ιούλιο και η Κομισιόν, ο Ζαν Κλοντ κάνει μια έκκληση σε όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να αναλάβουν τις ευθύνες τους επί τη βάση της προτάσεως της Κομισιόν με την ισχυρή υποστήριξη του Κοινοβουλίου. Τώρα εξ ονόματος του Συμβουλίου το λόγο έχει η κυρία Καλνίνα Λουκατσέβικα. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση. Πρώτα για τη μετανάστευση. Όπως είπα ήδη, το Συμβούλιο προσπαθεί να πετύχει μια καλή ισορροπία για μακροπρόθεσμες λύσεις. Καταλαβαίνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εμείνει στην πρότασή της. Το Συμβούλιο όμως δεν είναι πεπισμένο ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να λυθούν οι αιτίε του προβλήματος και όχι να καταπολεμήσουμε μόνο ε, τα συμπτώματα. Αξιότιμοι ευρωβουλευτές, αν έχουμε πλημμύρες επανειλημμένος, πρέπει να φτιάξουμε ένα φράγμα. Και επιτρέψτε μου να επαναλάβω αυτό που είπα και στην αρχή. Κανείς στο Συμβούλιο δεν αμφισβητεί το γεγονός ότι πρέπει να βοηθήσουμε αυτούς που πραγματικά χρειάζονται βοήθεια. Κανείς δεν αμφισβητεί την ανάγκη να ενισχύσουμε την αναπτυξιακή μας συνεργασία. Κανείς δεν αμφισβητεί τη συνεργασία με τις και τις χώρες transit. Όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα των παράνομων διακινητών. Αλλά πρέπει να συζητήσουμε για να βρούμε ποια είναι η καλύτερη δυνατόν λύση. Πρέπει να βρούμε μια μακροπρόθεσμη λύση, μια λύση που να φέρνει αποτελέσματα. Συγχρόνως το Συμβούλιο πάντα ήταν έτοιμο να αντιδράσει. Έχουμε δουλέψει δραστήρια και τον Απρίλιο προκειμένου να βρεθεί κάποια λύση και να αποφύγουμε να χάνονται τόσες ζωές στη Μεσόγειο. Τριπλασιάσαμε τον προπολογισμό της Frontex. Οι χώρες μέλη έδωσαν επιπλέον τεχνικά μέσα για να βοηθήσουν την Frontex, κάτι το οποίο βοήθησε να σωθούν ζωές στην Μεσόγειο και να μην επαναληφθούν οι γνωστές τραγωδίες τον Απριλίο. Όπως είπα, το Συμβούλιο συμφώνησε επίσης για δράση στην Μεσόγειο στα πλαίσια της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Το Συμβούλιο επίσης ενισχύει τη συνεργασία του με τις χώρες προέλευσης και τις χώρες transit από όπου περνούν οι πρόσφυγες. Θέλει να βρει μια συνολική λύση το Συμβούλιο στον τομέα της μετανάστευσης. Έρχομαι στην Ελλάδα τώρα. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ανυπομονησία από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όλοι έχουμε τα μάτια στραμμένα στην Ελλάδα και όλοι καταλαβαίνουμε και συμφωνώ και εγώ ότι δεν είναι απλή κατάσταση. Όμως πρέπει να επιτρέψουμε στην Ελλάδα να δείξει σε όλους μας ότι είναι σε θέση να προσφέρει ένα σχέδιο μεταρρυθμίσεων και ότι είναι σε θέση να το θέσει και σε εφαρμογή. Η αυριανή διάσκεψη, ελπίζω, θα φέρει θετικά αποτελέσματα. Κανείς δεν πνίγεται επειδή πέφτει στο νερό, αλλά επειδή παραμένει στο νερό για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Θέλουμε να βοηθήσουμε την Ελλάδα να βγει από το νερό. Οι μεταρρυθμίσεις πολλές φορές πονάνε. Αλλά ακόμα και από την εμπειρία που έχω εγώ στη χώρα μου, μπορώ να σας πω ότι οι άνθρωποι εκτιμούν την πολυπλοκότητα των αποφάσεων της κυβέρνησης που είναι σκληρές οι αποφάσεις αυτές, αλλά χρειάζονται, χρειάζεται μια λύση και όχι μια συνεχιζόμενη ε, αγωνία ή μια στάσιμη κατάσταση. Χρειαζόμαστε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που να είναι δυνατή, ευημερούσα. Θέλουμε μια ενωμένη ευρωπαϊκή οικονομία. Γι' αυτό πρέπει να ξεπεράσουμε τα εμπόδια πρέπει να δράσουμε με θάρρος. Πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Η ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου συμπεριλαμβάνει και πολλά θέματα που έχουν να κάνουν με την οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την έκθεση των πέντε προέδρων, τις αναχώρασης τάσης και την ενίσχυση της ασφάλειας στο εσωτερικό και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά τα θέματα είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση που είχαμε εδώ σήμερα και επιτρέψτε μου να υποφελθώ από την ευκαιρία για να σας ευχαριστήσω από βάθους καρδίας για την καρποφόρα συνεργασία που είχαμε το εξάμεινο της Λετωνικής Προεδρίας. Οι συζητήσεις μας ήταν πολύ ενδιαφέρουσες, γεμάτες δυναμισμό. Προσπαθήσαμε να βρούμε λύσεις παρά τα δύσκολα θέματα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Η συνένεση είναι κάτι πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν και προς την ε, Νέα Λουξεμβουργιανή Προεδρία και προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλω να πω ότι ελπίζω να είναι περισσότερο ειρηνική επόμενη έξι μήνες με περισσότερη ανάπτυξη και ευημερία. Ευχαριστώ. Και το Κοινοβούλιο ευχαριστεί την ε, απερχόμενη Προεδρία για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε στη διάρκεια των περασμένων έξι μηνών. Σας ευχαριστώ και πάλι και εδώ τελειώνει η συζήτηση αυτή. Da, continuăm uh, συνεχίσουμε με την ε, έκθεση. Προηγουμένως όμως υπάρχει μια αίτηση παρέμβασης από τον κύριο Γλέζο. Για διαδικαστικό θέμα. Κύριε Γλέζο, έχετε το λόγο. Ε, δεν ζήτησα λόγο για διαδικαστικό θέμα. Ζήτησα το λόγο για την προηγούμενη συζήτηση μου υποσχέθηκε το Προεδρείο ότι θα μου το δώσει και δεν μου τον έδωσε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και θέλω, ζήτησα ένα λεπτό να μιλήσω στο προηγούμενο θέμα. Μου είπε ναι, μου έστειλε εκπρόσωπο να μιλήσω και τελικά δεν μου έδωσε το λόγο. Τι να κάνω τώρα εγώ. την am Από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Γλέζο, το πρόβλημα είναι ότι η προηγούμενη συζήτηση ήταν απλώς μια συζήτηση για τους επικεφαλείς των πολιτικών ομάδων. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι κανένα άλλο μέλος δεν έχει το δικαίωμα να λάβει το λόγο. Αν υπήρχε κάποια δυνατότητα, θα είχατε τη δυνατότητα να λάβετε το λόγο και να μιλήσετε, λέει ο πρόεδρος. Αλλά τώρα, τώρα μπορείτε να λάβετε το λόγο. Τώρα. Yes. Μπορείτε να μιλήσετε τώρα. Θέλω να θέσω και ήθελα να θέσω ένα ερώτημα σε όλους τους συναδέλφους. Ένα ερώτημα το οποίο θεωρώ κέριο για την πορεία της Ευρώπης αν θέλει να είναι δημοκρατική. Το ερώτημα είναι θα σεβαστούμε τη βούληση ενός λαού ναι ή όχι. Ο ελληνικός λαός αποφάσισε με τις εκλογές ότι δεν θέλει δάνεια, δεν θέλει αυτό την πορεία θέλει τη δική του να φτιάξει το δικό του μέλλον. Θα το σεβαστούμε ναι ή όχι. Δεν είναι θέμα του ελληνικού λαού, είναι θέμα δημοκρατίας. Θα σεβόμαστε τη βούληση ενός λαού όποιου και αν είναι ναι ή όχι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ο ελληνικός λαός αποφάσισε και οικοδομεί το παρόν και το μέλλον του και δεν θέλει να τον πνίξουν οι δανειστές του. Οι διαπραγματεύσεις δεν οδήγησαν πουθενά. Μία λύση μονάχα υπήρχε. Ούτε ρήξη, ούτε υποταγή. Μετά από ένα χρόνο ελάτε να συζητήσουμε. Και αν χρωστάμε να τα πληρώσουμε. Αν δεν χρωστάμε να μην πληρώσουμε. Αυτό ήθελα να πω και παρακαλώ επειδή φεύγω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε 20 μέρες θέλω το ερώτημα αυτό ο κάθε βουλευτής να απαντήσει με τη συνείδησή του και να ξέρετε θα σας κυνηγάει η άποψή μου όπου και αν πάτε και όπου και αν πάω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γλέζο. Προχωρούμε στο επόμενο σημείο της σημερινής της διάταξης. Πρόκειται για την έκθεση του κυρίου Φερνάντες και του κυρίου Μπούλμαν